Επανέναρξη της συνεδρίασης. Και τώρα έχουμε την δήλωση της είπα, της εκπρόσωπου για θέματα πολιτικής ε, ασφαλείας και εξωτερικής πολιτικής για την ε, κατάσταση στην Ουκρανία. Κύριε Επίτροπε, έχει το λόγο.